Dear let's start this uh, joint... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε με την κοινή συνεδρίαση ε, των Επιτροπών ΑΦΚΟ και ε, ΕΚΟΝ. Θα συμπροεδρεύσω με την πρόεδρο της ΑΦΚΟ θα υιοθετήσουμε στην αρχή την ημερήσια διάταξη και πρέπει επίσης να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 20ης ε, ε, Μαρτίου. Δεν έχουμε κάποιες ε, ανακοινώσεις. το ζήτημα της συνάντησης αφορά την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι, ε, ποια είναι η βάση αυτής της συζήτησης, ε, το ε, Brexit και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι κατευθείαν μπορώ να δώσω τον λόγο ε, στον Δανούτα ε, ε, για να, στην Δανούτα για να δώσει μία πρώτη επεξήγηση μαζί με τον κύριο Μάτο. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ως ε, Πρόεδρος θα ήθελα να σας θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα εξαιτία της ανάγκης τροποποίησης ε, του άρθρου 22 ύστερα από την απόφαση του δικαστηρίου του 2011 ε, όπου υπήρχε μια υπόθεση μεταξύ Ηνωμένου Βουσιλείου κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και γι' αυτό το λόγο εργαζόμαστε ε, πάνω σε αυτή την έκθεση που, θα, ε, αφορά την αλλαγή ε, του άρθρου έχει σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και θα ε, δώσει τη δυνατότητα στο, ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα να έχει εξουσία όσον αφορά τα CCP. Στην συνέχεια θα μιλήσει και ο συνάδελφος. Έχουμε προτείνει τρεις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις καθώς επίσης και στο καταστατικό. Όπως ε, γνωρίζετε, στην περίπτωση των CCP έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν, ε, ε, έναν τομέα όπου ε, υπάρχει η δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τους νομοθέτες, όμως υπάρχει ο κίνδυνος και, το, και η Κεντρική Τράπεζα να, να παρεμβαίνει και έτσι λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε παράλληλες αποφάσεις οι οποίες θα αλληλεπικαλύπτονται και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να θέλουμε θέσουμε ένα πλαίσιο με την τροπολογία 4 ε, σχετικά ε, σχετικά με τις ε, πιο συγκεκριμένες δικαιοδοσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα CCP και θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 22 όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών όμως τα συστήματα κανονισμών έχουμε τα συστήματα συμψηφισμών και ε, πληρωμών τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, με έναν τρόπο ο οποίος θα, σε, θα σέβεται ε, την νομική πράξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να εφαρμόσουν τέτοιες πράξεις και επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σκοπεύουμε επίσης Αναλογιζόμαστε επίσης και σχεδιαζούμε ε, τροπολογίες ε, για να αντικαταστήσουν την έννοια της αναγνώρισης. Ε, δεν ξέρω αν ε, σκέφτεστε και εσείς το παρόμοιο. Ε, αυτό είναι το πρώτο μου σημείο, να δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό το πλαίσιο για τα CCP σχετικά με το ποιος έχει το δικαίωμα να νομοθετεί και επίσης να σεβόμαστε τις εξουσίες των διαφόρων θεσμών. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω αφορά ε, τα όρια μεταξύ αυτού του φακέλου και του φακέλου για το ΕΜΙΡ και εδώ θα ήθελα ε, να πω ότι το άρθρο 22 ε, του καταστατικού ορίζει τι ε, μπορεί να κάνει το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς επίσης και άλλες κεντρικές τράπεζες όσον αφορά τα CCP ε, και, αυτός, ε, και αυτό είναι το Lex Generalis το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα για τροπολογίας ε, η διατύπωση είναι αρκετά ευρύ, ώστε να καλύπτει όλα τα περιστατικά ε, και οτιδήποτε και αν προκύψει ότι ε, περιορισμοί και αν εμφανιστούν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσουμε να το συμπεριλάβουμε στο καταστατικό και θα περιορίζουν αυτή την εξουσία και γι' αυτό το λόγο δεν το κάνουμε όσον αφορά το καταστατικό. Η επιλογή λοιπόν που κάναμε ήταν να αφήσουμε ε, την διατύπωση ως έχει ε, για να είναι όσο ε, ευρία όσο ήταν και στην αρχική πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα. Επίσης προσθέτουμε τον περιορισμό όσον αφορά τον, τον σεβασμό των εξουσιών των συνομοθετών και ως ε, συνομοθέτης θεωρούμε ότι οι εξουσίες μας θα πρέπει ε, να αναγνωρίζονται και να σέβονται. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει την ελευθερία να ε, δρά σε έκτα, περιπτώσεις εκτακτών αναγκών, όπως προβλέπεται και από τον κανονισμό ΕΜΗΡ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να λάβει μέτρα με βάση ε, αυτό για να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση ε, που τα CCP δημιουργούν εντάσεις ε, στην αγορά όσον αφορά την νομισματική πολιτική και αυτό συσχετίζεται με το ΕΜΗΡ και αυτή η επιλογή ευελιξίας έχει να κάνει με τη δυνατότητα του Εμμύρ να ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, όσον αφορά τα CCP ε, και την αναγνώριση των CCP και το τελευταίο σημείο αφορά το ότι εισάγαμε μια αιτιολογική σκέψη σχετικά με ε, το καταστατικό που ορίζουν προϋποθέσεις ε, ε, όπου η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει ε, να επιβάλλει και αυτό φαίνεται στην τροπολογία 2 της 8ης αιτιολογικής σκέψης. Ε, έχουμε ανοιχτή τη λίστα αυτής της αιτιολογικής σκέψης ούτως ώστε το καταστατικό να, έχει, να είναι αρκετά ευρύ και ανοιχτό ε, κάτι το οποίο επιθυμούμε για έναν ε, θεσμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ε, πιστεύουμε ότι αυτό χρειάζεται σε αυτήν την ιδεολογική σκέψη διότι έχει ως στόχο να κατευθύνει μελλοντικές ερμηνείες του κειμένου και σε μελλοντικές υποθέσεις που μπορεί να προκύψουν ώστε να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον οι εξουσίες που δίνονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά την, τα CCP θα μπορούν να εφαρμόζεται. Αυτό είναι το νόημα και η νομική διαδικασία που εφαρμόζουμε εδώ πέρα ε, για ούτως ώστε όλα να είναι ξεκάθαρα και χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάσουμε τον κανονισμό που είναι αναγκαίος για τον καταστατικό και για να ε, περιορίσουμε και δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ε, ε, εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά η αιτιολογική σκέψη αποσκοπεί στο να είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα τα οποία αφορούν και τον ΕΜΗΡ. Αυτά λίγο πολύ σχετικά με τη συγκεκριμένη προσέγγιση καθώς επίσης και όσον αφορά την διατύπωση που έχουμε ε, προτείνει για το άρθρο 22. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο συνεισηγητής από την εικόνα, ο Γκαμπριέλ Μάτορ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έλεγε η συνάδελφος ότι θα συμπληρώσω την παρουσίασή της. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όμως ήταν αρκετά ε, εμπεριστατωμένη. Δύο πράγματα, δύο αποχρώσεις. Καταρχάς να ευχαριστήσω και την ίδια και την ομάδα της ε, για την ευκολία με την οποία συνεργαστήκαμε και επίσης να πω ότι χαίρομαι που μπορούμε να τηρήσουμε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ώστε να τελειώσουμε πριν από το καλοκαίρι. Βεβαίω ε, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να πω ότι μου φαίνεται αδιανόητο ότι ακόμα δεν έχουμε τη νομική γνωμοδότηση που έχουμε ζητήσει. Επισήμω μάλιστα τον Ιανουάριο και ε, άτυπα από τον Οκτώβριο. Αποφασίσαμε λοιπόν οι δύο συνεισηγητές σε αυτή την περίπτωση να συνεχίσουμε ε, να υποστηρίζουμε την πρότασή μας για να μην καθυστερήσουμε κι άλλο αυτή την πρόταση και να μην ε, υπάρχει και πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα. Πολύ σύντομα να πω ότι πιστεύω ότι ο στόχος αυτής της πρότασης είναι σαφής. Ε, να υπάρχουν αυτές οι νομοθετικές αρμοδιότητες ώστε να υπάρχουν δεσμευτικές ε, συνθήκες και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους σε στενή συνεργασία με άλλους ε, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, δεχόμαστε με ικανοποίηση την πρόταση που είχε γίνει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα όσον αφορά ε, τη δημιουργία ενός πραγματικού συστήματος εποπτείας ε, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και φυσικά να υπάρχει και αντίστοιχη ε, θετική επιρροή για τις κεντρικές τράπεζες. Όλα αυτά βέβαια πλαισιώνονται από την ανάγκη να γίνει σεβαστό το θέμα των αρμοδιοτήτων λαμβάνοντα υπόψη ποιε υπηρεσίε και όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να καθορίσουν το ε, πλαίσιο που αφορά το κεντρικό τη συμβαλόμενο. Και φυσικά οι νέε αρμοδιότητε ε, τη ΕΚΤ βάσει του άρθρου 22 ε, που σημαίνει ότι πρέπει να έρχεται σε επαφή υποχρεωτικά και με άλλου οργανισμού. Το είπε η συνάδελφο Χούμπνερ για ε, νόμους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας ε, στις αιτιολογικές σκέψεις έχουμε συμπεριλάβει ε, ένα κατάλογο αρμοδιοτήτων σε αυτή την διορθωτική πράξη και πιστεύουμε ότι το πιο λογικό είναι να είναι ανοιχτός αυτός ο κατάλογος, να μην κλείσει. Γι' αυτό ακριβώς και κάναμε και την πρόταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα να πούμε πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει σε κάθε έκτακτη περίσταση η ΕΚΤ και έχουμε περιλάβει όλες τις ε, πιθανές συνθήκες. Ελπίζω να γίνει αποδεκτή η πρόταση και ε, πολύ ευχαριστώ να τη συζητήσουμε με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και τους υπόλοιπους ε, σκιώδης ηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Περνάμε στους σκιώδης ηγητές και από ΕΚΟΝ και από ε, ΑΦΚΟ η υπερβάνηση ευχαριστώ για τις προτάσεις αυτές. Θα επαναλάβω την παρατήρηση τη ηγητού από την ΕΚΟΝ, της ηγητρίας, από την ΕΚΟΝ. Πρόκειται για ένα τομέα που θέλουμε να ρυθμίσουμε τα νομικά ζητήματα. Είναι ένα τομέα όπου είμαστε συνομοθέτες, θέλουμε να λειτουργεί σωστά η νέα αγορά. και να είναι ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Θέσαμε λοιπόν και μια σειρά από στην νομική υπηρεσία. Αν δεν έχουμε τις απαντήσεις δεν νομίζω ότι μπορούν να προχωρήσουν οι δύο συγητές. Δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές. Είτε έκτο το Συμβούλιο ως βασικό στόχο έχουν ουσιαστικά να ξεμπλοκάρουν τα πράγματα και να δουν πώς μπορούμε να βρούμε μια διέξοδο. Να γίνει σεβαστό το χρονοδιάγραμμα, δεν έχω αντίρρηση, αλλά είναι γελίο να προχωρούμε. Και λέτε κιόλα ε, ποια είναι η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών χωρίς να έχουμε λάβει την ε, νομική γνωμάτευση. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Επί της ουσία για τις τροπολογίες. απλουστευμένη διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού της ΕΚΤ για να προχωρήσουμε σε αυτό το χρόνο. Παράλληλα εγκρίνουμε και την νομοθεσία ημίρ 2.2 για την πρώτη τροπολογία που είναι διευκρινιστικής φύσεως για να δούμε ε, τη διατύπωση τώρα ακριβώς. Εντάξει, πάντως δεν έχω πρόβλημα για τις άλλες δύο τροπολογίες Άκουσα με προσοχή και διαβάζω ότι λέει και για τις δύο περιπτώσεις ότι δεν έχουμε πλήρης εξαντλητικούς καταλόγους αποκλειστικούς but not limited to, μάλιστα, διευκρινίζει η δεύτερη τροπολογία. Χρειάζεται όμως, σίγουρα, ο κατάλογος αυτός. Πρέπει να το δούμε, να το επαληθεύσουμε. Κομισιόν η Κεντρική Τράπεζα εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Καλό θα ήταν, αν είναι, να πάρουν το λόγο. Και για την τροπολογία, για το καταστατικό αυτό καθεαυτό, καταλαβαίνω ότι επιδιώκουν οι δύο συνεισηγητές. Αντί να κινήσουν από την πρόταση της ΕΚΤ, εμπνεύστηκαν από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που και αυτή όμως για μένα είναι προβληματική. Πρέπει λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Θα διευρύνουμε γενικά την εντολή της ΕΚΤ, όπως προτείνει η ίδια. Παρότι ασκήθηκαν κριτικές ότι ίσως είναι πολύ ευρεία η εντολή και ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σηματότητας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά τροπολογία. Και εκεί είναι σημαντικό να μας απαντήσει η νομική υπηρεσία. Πρέπει να πούμε στην ΕΚΤ, πρέπει να σεβαστείτε την δευτερογενή νομοθεσία για την εκπλήρωση των καθηκόντων σας. Η διατύπωση που μας προτείνει ο συνεισηγητής, που δεν είναι ακριβώς η ίδια διατύπωση με αυτή που προτείνει η Κομισιόν, κοντά είναι βέβαια. Τι λέει η Κομισιόν για να δω εκεί. Προτείνει consistent η Κομισιόν. Εδώ λέμε full respect, I recognize. Αλλά η λογική παραμένει ίδια. Προς τα εκεί θέλουμε να οδεύσουμε. Εγώ δεν μπορώ να αποφανθώ. Προς το παρόν τουλάχιστον. Πρώτα, σε ευχαριστώ. ECR, Μπεντ Λούκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τους δύο σκιώδεις εισηγητές, την Σάντρα Λούνες και τον Μόρτεν Μέσσερ Σμιτ, που ζητούν συγγνώμη. Δεν μπορούν να είναι εδώ. Έχουν προετοιμάσει πάρα πολύ σύντομα σημειώματα ε, που θα τα διαβάσω εξ ονόματός τους. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές για την έκθεση Συζητούμε την πρόταση αυτή διότι υπάρχει νομική ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 22 του καταστατικού της ΕΚΤΑ και του συστήματος κεντρικών τραπεζών για νομισματικούς σκοπούς θέλουμε να διευρύνουμε την εντολή της ΕΚΤ. Το σχέδιο έκθεσης προτείνει ευπρόσδεκτες τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν η ΕΣΥΑΡ θα καταθέσει τροπολογίες ώστε ΕΚΤ να μπορεί να φέρει σε πέρα απαιτήσει στο ΕΜΙΡ και τη σχετική νομοθεσία χωρίς να δίνουμε όμως βέβαια και εν λευκό εξουσιοδότηση στην ΕΚΤ. Αυτά, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ ο Πρόεδρος. Κύριο Γέζεκ Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του συνεισηγητέ για το σχέδιο έκθεση. Στηρίζουμε και εμεί το στόχο των τροπολογιών που κατέθεσε η ΕΚΤΑ. Συμφωνώ όμως με την Κομισιόν ότι αυτές οι αρμοδιότητες, οι διευρυμένες θα πρέπει να πλαισιωθούν σωστά στο πλαίσιο της τάμης νομοθεσίας. Οι, οι δηλαδή πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους. Έχουμε τις τροπολογίες των συνεισηγητών και τις προτάσεις τους να γίνει σεβαστή πλήρωση σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Καταλαβαίνω τη θέση αυτή, όμως έχω κάποιες ανησυχίες Μήπως δεν δοθεί η επαρκή ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να φέρει σε πέραση τα βασικά της καθήκοντα από άπτονται της νομισματικής πολιτικής. Και αυτό θα ισχύσει ιδίω, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, σε απρόβλεπτες καταστάσεις και συμβάντα που μπορεί να μην καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης περιορισμός εντολής ε, της ΕΚΤ και των εξουσιών σημαίνει ότι δεν θα μπορεί ανεξάρτητα να αναλάβει δράση σε τέτοια περίπτωση. Αν έχουμε δηλαδή ένα συστημικό συμβάν για που απειλεί την νομισματική σταθερότητα τη Ένωση, Διότι περιορίζεται και πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρω με τη νομοθεσία τη Ένωση. Η ΕΚΤ και δεν μπορεί να δράσει στο πνεύμα αυτή των συνθήκων και τη νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι καλό θα ήταν ίσως να επανέλθουμε σε μια πιο ευρεία διατύπωση σύμφωνα με τις προτάσεις της Κομισιόν. Ε, ότι δηλαδή οι ρυθμιστές, οι κανονισμοί μάλλον που προτείνει η ΕΚΤ θα πρέπει να συνάδουν consistent with με τις προτάσεις των συνομοθετών. Υπάρχει υποστήριξη για αλλαγή του καταστατικού της ΕΚΤ για να μπορεί να φέρει σε πέρας καθήκοντα που είναι ζωτικά για την σταθερότητα της Ένωσης. Όχι μόνο τα επόμενα χρόνια, αλλά μακροπρόθεσμα. Οι περιορισμοί ε, των ορμοδιοτήτων και εξουσιών κατέστασαν σαφείς ε, στην απόφαση του δικαστήριου του 2015 που ε, επιβάλλει και τις αλλαγές. Ο καταστατικό ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σβέν Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για το έργο τους. Γενικά συμφωνούμε με την ανάγκη να ξεκαθαριστεί ότι έχει τις εξουσίες αυτές η ΕΚΤ και στην Ένωση και απέναντι σε τρίτες χώρες κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για να γίνουν και ιδέωσες αλλαγές. Πιστεύουμε βέβαια ότι στη διατύπωση θα πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι και σαφείς. Να υπάρχει δηλαδή πλήρη συνέπεια με το γενικό νομοθετικό πλαίσιο. Σε κάποιες λεπτομέρειες η διατύπωση δεν οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα προς το παρόν και συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που είπε περές επ' αυτού. Δηλαδή μέχρι στιγμής λέει θα πρέπει να σέβεται, it should respect, στο άρθρο 5. Δεν είναι το ίδιο με το fully consistent, να συνάδει πλήρω. Καταλαβαίνω ότι εκτ και άκουσα και αυτό που είπατε Πιέτρ όλοι και η ΕΚΤ φυσικά θα ήθελε να έχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά αν δίνεται αυτή η ευελιξία θα πρέπει να κατοχυρώνεται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς, δεν ξέρω. Αν αυτό καταστεί αναγκαίο θα πρέπει να εκχωρηθεί από τους συνομοθέτες και όχι με μια γενική τέτοια ρήτρα. Θέλω να ακούσω τι λέει όμως και η Κομισιόν και η ΕΚΤ σε σχέση με τις προτάσεις. Μα θέλω να ακούσω και την άποψη της ΕΚΤΑ για την έκθεση της Κομισιόν και για το έργο των συνεισηγητών. Ευχαριστώ. Uh, Ο κύριος Πιέργας, ο κύριος Κοστάλντο δεν είναι εδώ. Κύριε Μοντρό. κανείς. Οπότε με ναι, catch the eye. Ωραία, έχουμε την ε, Κομισιόν. Καθώς επίσης και εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ξέρω αν θα θέλετε το λόγο. Κανονικά δίνουμε το λόγο στην ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πιστεύω ότι ε, όπως υπόθηκε και ε, στην, προηγούμενη ε, συζήτηση οι τροπολογίες για το άρθρο 22 είναι σημαντικά για να επιτρέψουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να κάνει το έργο της όσον αφορά την αναγνώριση και την επίβληψη των CCP. Και γι' αυτό το λόγο καλωσορίζουμε τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να προχωρήσει ο συγκεκριμένος ε, φάκελος όσον αφορά τώρα την ουσία. Ε, χαιρετίζουμε τους εισηγητές ε, και την υποστήριξή τους για την τροπολογία του καταστατικού, του άρθρου 22 του καταστατικού και επίσης την συνοχή που υπάρχει σχετικά με την λήψη μελλοντικών αποφάσεων Όσον αφορά τα ε, ζητήματα της ε, διατύπωσης θα επανέλθουμε σε μελλοντική στιγμή. Δεν ξέρω αν ο κύριος ε, Μαρμαράς θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Θα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στείλει κάποιον να ε, συμμετάσχει στη συζήτηση. Ο κύριο Σνάτο Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις. Για την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πω ότι συμφωνώ μαζί της πρέπει να έχουμε το συντομότερο δυνατόν μια νομική γνωμοδότηση η οποία έχει καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο πάνω από πέντε μήνες ε, και νομίζω ότι μπορούμε να τα τροποποιήσουμε και ανάλογα με τα όσα θα λένε οι ε, συστάσεις εκεί. Όσον αφορά τον ανοιχτό κατάλογο, προσωπικά πιστεύω ότι η πρόταση ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη ε, σαφήνεια στην ερμηνεία. Δεν θα κλείσει να παραμείνει ανοιχτός για να προσθεθεί οτιδήποτε θεωρηθεί απαραίτητο. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι δίνουμε λευκή επιταγή στην ΕΚΤ. Νομίζω ότι αυτό το είπαμε και δεν θα έπρεπε να ανησυχεί κανένα κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την ερμηνεία του κυρίου Γιάτσεκ, ε, κοιτάξτε. Εγώ νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ένας κάποιος περιορισμός, αλλά λογικά σεβόμενοι την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κυρίως επιτρέποντας να μπορέσει να τηρήσει τους στόχους της νομισματικής πολιτικής που είναι από τους βασικούς τους ε, στόχους. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε κάλλιστα σε ένα κείμενο στο οποίο θα συμφωνούμε όλοι και δεν θα έχει προβλήματα. Και νομίζω ότι σε αυτό στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε πλήρως τις αρμοδιότητες του κάθε οργάνου. Επομένω πρέπει να εργαστούμε προ αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά ειλικρινά πιστεύω ότι έτσι όπω έχει τεθεί η έκθεση ε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε παρατήρηση. Ευχαριστώ. Η Ντανούτα, μπορεί να μιλήσει στη συνέχεια. Η πρότασή σου για αυτή την αιτιολογική σκέψη που όπως είπες είναι πολύ σημαντική Υπάρχει μια ερώτηση από την ΕΚΟΝ προ την ΑΦΚΟ. Οι αιτιολογικέ σκέψει είναι σημαντικέ για την νομοθεσία και σε αυτή την περίπτωση, αλλά αυτή δεν είναι αιτιολογική σκέψη συγκεκριμένη, είναι αιτιολογική σκέψη για το καταστατικό, που δεν θα συμπεριληφθεί δηλαδή στο καταστατικό. Είναι μια αιτιολογική σκέψη του κειμένου τη συναπόφαση που τροποποιεί το καταστατικό, αλλά δεν έχει την έννοια που έχει μια αιτιολογική σκέψη ενό κανονισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν το έχετε σκεφτεί αυτό και αν έχετε λάβει υπόψη τι νομική επίδραση έχει αυτή η αιτιολογική σκέψη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με τη διατύπωση αυτή. Αναφερόμαστε στο, άρθρο. αφήνω, στο άρθρο. Αφήνω την αιτιολογική σκέψη που είναι δεύτερο ζήτημα να μιλήσω για το άρθρο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαμε τον όρο consistent. Η ανταλλαγή απόψεων που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, μας ε, έδειξε ότι δεν τους άρεσε ο όρος consistent και θα προτιμούσαν να έχουν μια φράση του τύπου taking into account. Για μας είπαμε ότι είναι περισσότερο από αυτό, διότι ο όρος respecting ε, θα μπορούσαν να θεωρήσουν κάτι ότι ξεκινάει μια ιεραρχία μια ιεράρχηση. Εμεί θέλαμε κάτι που να αντανακλά την πραγματικότητα, να μην υπάρχει ιεράρχηση, γιατί δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει ιεράρχηση και ε, να σημαίνει πολύ περισσότερο από το take into account. Γι' αυτό ακριβώ ε, εξακολουθώ να σκέφτομαι και να προβληματίζομαι από αυτού ε, και εχθέ ε, ρώτησα και του συναδέλφου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά πόσον ο όρο recognize αντί για respect θα ήταν αποδεκτό και από ό,τι κατάλαβα ε, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ ε, τον δέχεται. Αν κάποιος έχει κάποια καλύτερη πρόταση από το Recognize, πολύ ευχαρίστω να την ακούσουμε, αλλά να σας πω ότι ψάχνουμε έναν όρο που να είναι αρκετά ισχυρός και ταυτόχρονα να ε, υποχρεώνει την ΕΚΤ να σέβεται και να λαμβάνει υπόψη της το ρόλο του συνομοθέτη, αλλά εγώ προσωπικά πίστευα ότι το take into account δεν αρκεί. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το recognize και να λέμε ότι αναγνωρίζει πλήρως το ρόλο του συνομοθέτη. Θεώρησα ότι ήταν καλύτερο. Έχουμε χρόνο για τροπολογίες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι αυτή η διατύπωση χρησιμοποιήθηκε στη συζήτηση μέχρι τώρα και μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα το βρούμε. Δεν είναι και τεράστια αλλαγή. Πρώτο αυτό λοιπόν. Δεύτερον, όπως προσπάθησα να εξηγήσω και στην εισαγωγή μου, δεν μπορούσαμε στο καταστατικό να προσθέσουμε οποιονδήποτε κατάλογο, ο οποίος τα περιορίζει την εξουσία δράσης της ΣΕΚΤ. Αλλά θέλαμε να υπάρχει αναφορά στον κατάλογο των πιθανών δράσεων, διότι θεωρούμε ότι αυτό δείχνει την πρόταση του νομοθέτη. Αν ε, στο μέλλον υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος θα προσφύγει και πάλι στο δικαστήριο, τα θέματα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Αυτή λοιπόν είναι η πρόθεσή μας. Εάν ε, λάβουμε και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, ε, η οποία μπορεί να προτείνει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, τότε σίγουρα μπορούμε να το λάβουμε υπόψη αλλά νομίζω ότι δεδομένη της σημασίας των ε, θεμάτων αυτών, που είναι ο πιθανός αντίκτυπος ε, στη νομισματική πολιτική, επιλέξαμε να αφήσουμε τη διατύπωση του καταστατικού ουσιαστικά αυτούσια, όπως την πρότεινε η ΕΚΤ. Με μόνη αλλαγή, αυτή την ανάγκη να γίνονται σεβαστέ οι εξουσίες ε, του συνομοθέτη. Ε, κατά τα άλλα έχουμε τη διατύπωση της ΕΚΤ και μετά έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει it should be consistent, να υπάρχει συνέπεια με το συνομοθέτη. Εμείς λέμε recognize, ε, αλλά η ΕΚΤ η ίδια ήταν αυτή η οποία πρότεινε τη συγκεκριμένη διατύπωση που δεν περιορίζει τις εξουσίες τους και ταυτόχρονα τους δίνει και το ελεύθερο να δράσουν σε κατεπίγουσε περιπτώσεις και να λάβουν μέτρα τα οποία μπορεί να χρειαστούν σε αυτή την περίπτωση. Αυτή, αυτό είναι το όλο σκεπτικό. Το αίτημα προ το συμπρόεδρο είναι το εξή. Επειδή τώρα πρέπει να αποφασίσουμε αν η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών όπως ε, προτείνουμε εμείς ε, είναι πριν λάβουμε την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε ως προθεσμία τη Δευτέρα Μαΐου, αλλά δεν μπορούμε, δεν να ξέρουμε πότε θα μας δώσει τα στοιχεία η νομική υπηρεσία. Έχετε δίκιο, δεν θέλω να ξανανοίξω τη συζήτηση, έχουμε πολύ χρόνο. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ακόμα δεν έχω πιστεί ότι έχουμε βρει τη σωστή διατύπωση και τη σωστή λύση. Είναι πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. και υπάρχει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει το κείμενο της ΕΚΤ, εγώ προσωπικά δεν έχω βρει πιστική λύση. Μπορεί και να μην υπάρχει, μπορεί να μην είναι δυνατόν. Μπορεί ε, ε, το πιο απλό να μην είχε αποφασιστεί όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο ε, και να ήταν έτσι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή τώρα υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να το τροποποιήσουμε, έχει γίνει πιο περίπλοκο. Για το λόγο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι επειδή έχουμε ζητήσει και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, θα πρέπει να δούμε και δεν έχει νόημα να, να πάρουμε τροπολογίες ε, πριν ε, ε, λάβουμε και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Πρέπει να δώσουμε μια προθεσμία που θα δίνει το χρόνο και στα μέλη να εξετάσουν και τη γνωμοδότηση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μια ε, επιπόλαιη γνωμοδότηση, είναι σημαντική. Σχόλιο εκτός μικροθόνου από τον κύριο Μπροκ. Μπορούμε να τα αφήσουμε ανοιχτό, να το ελέγξουμε με την νομική υπηρεσία, να ξέρουμε πότε θα τη λάβουμε αυτή τη γνωμοδότηση και να δώσουμε και αρκετό χρόνο τα μέλη. Yeah, exactly. So we will not be ε, δεν θα είναι δύο ώρες μετά τη γνωμοδότηση, προφανώς θα υπάρχει και χρόνος. Δώστε μας όμως λίγο χρόνο, δεν μπορούμε να σας πούμε τώρα. Θα το συζητήσουμε και με την νομική υπηρεσία και μεταξύ μας και θα σας διαβιβάσουμε την ημερομηνία. Δεν χρειάζεται να σας πω το χρονοδιάγραμμα γιατί εξαρτάται και από αυτό. Μπορούμε όμως να κλείσουμε τη συνεδρία. Συντανούτα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω όλους εκείνους που ήρθαν και να ευχαριστήσω και τον Ρομπέρτο που προείδρευσε με τόση αποτελεσματικότητα. Η προθεσμία για τις τροπολογίες εξαρτάται από τη γνωμοδότηση. Και δεσμευόμαστε φυσικά να μιλήσουμε και πάλι με την νομική υπηρεσία και να δούμε τι απέκεινε αυτή η γνωμοδότηση. Να ευχαριστήσω και όλους εκείνους που συμμετέχουν και είχαν και τον κόπο να έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Πέραση συνεδρίασης. negotiating coordinators and everything, you know? The meeting with Gersan. Yes, it's in Okay, so. Negotiating. Okay, so the meeting is closed. Uh, there will be an incoming. Πέρα συνεδρίαση, σε ένα τέταρτο συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών για αυτού που ξέρουν για την ισοδυναμία τρίτων χωρών.